αύριο και θα ψηφιστεί αύριο η πρόταση για τη σύνθεση αυτή τη Επιτροπή. Περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η δήλωση του Συμβουλίου και τη Κομισιόν για την έκθεση διεύρυνση για το Μαυροβούνιο. Και πάλι θα δώσω το λόγο στον κύριο Βάνεν από την πλευρά του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρία Φίλε, θα ήθελα να χαιρετήσω την υποστήριξη του Κοινοβουλίου στις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει για να προχωρήσουμε τη διαδικασία ένταξη του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδίω χαιρετίζω την ε, προσπάθεια του εισηγητή σας, του Charles Κάνοκ, για να υπάρξει πρόθεση αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει ευρεία δημόσια υποστήριξη για την ενσωμάτωση του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης εθνική συνένεση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων του Μαυροβουνίου. Χάρη σε όλα αυτά, η χώρα αυτή έχει εργαστεί συστηματικά σε μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων το Δεκέμβριο, το προηγούμενο Δεκέμβριο και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρέτησαν την αξιολόγηση της Κομισιόν ότι το Μαυροβούνιο έχει επιτύχει ικανοποιητικά αποτελέσματα, ιδίω σε σχέση με τις κύριε προτεραιότητε που είχε θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010. Για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις ε, ένταξης τον Ιούνιο αυτού του έτους, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από το Συμβούλιο να εξετάσει την πρόοδο του Μαυροβουνίου στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αυτών. Μεταξύ αυτών είναι η πρόοδος στο κράτος δικαίου, ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα, ο αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματο και τη διαφθορά. Η Κομισιόν προετοιμάζει τώρα μια έκθεση για την εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων που θα παρουσιαστεί ενώπιον του Συμβουλίου κατά πάσα πιθανότητα το Μάιο. Το Μαυροβούνιο επέτυχε υψηλό επίπεδο εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξη και έχει προχωρήσει σημαντικά στην επίτευξη μια οικονομία τη αγορά και έχει προχωρήσει ιδιαίτερα στην βάση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Εταιρικής Σχέσης. Οι σχέσεις του Μαυροβουνίου με τους γειτονέ του είναι πολύ καλές και έχει εμπλακεί σε μια σειρά περιφερειακών πρωτοβουλειών, όπως η διαδικασία συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που, τις οποίες προείδευσε το Μαυροβούνιο το 2010 και 2011. Επίσης έχει εμπλακεί ιδιαίτερα στη διαδικασία του Σεράγεβο για την επίτευξη μιας λύσης για τους πρόσφυγες και τους εσωτερικά εκτοπισμένους στο Μαυροβούνιο, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Σερβία και Κροατία μετά από την σύγκρουση στην πρώην Ιουκοσλαβία στη δεκαετία του 1990. Αλλά έχει ακόμα δρόμο να διατρέξει το Μαυροβούνιο. Θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές του και να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Στον τομέα αυτό η πρόοδος είναι απαραίτητη Ιδίω σε σχέση με τα άτομα τα οποία είναι εκτοπισμένα μέσα στη χώρα του, την ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωση, την εφαρμογή πολιτικών κατά των διακρίσεων και τη ανεξαρτησία των δικαστικών. Προβλέπουμε στα συμπεράσματα της ε, συνταγματική μεταρρύθμισης που θα ενισχύσει την ανεξαρτησία τη δικαστική εξουσία Ο αγώνα κατά τη διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματο, θα είναι επίση σημαντικό για να προωθηθεί η πορεία του Μαυροβουνίου προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι πεπισμένο ότι θα επιτευχθεί πρόοδο. τη περιοχές αυτές και η διαδικασία ένταξης του Μαυροβουνίου θα δώσει μια περαιτέρω θετική όθηση στα Δυτικά Βαλκάνια. Με την ιστορική συμφωνία μεταξύ Πρίστινα και Βελιγραδίων και τη, η απόφαση να γίνει η Σερβία υποψήφια χώρα από την 1η ε, Μαρτίου του 2012 και με την πορεία της Κροατία που θα γίνει μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. υπάρχουν ισχυρά μηνύματα προ τι χώρε τη περιοχή που πρέπει να κάνουν τι απαραίτητε πολιτικέ επιλογέ για να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στα πλαίσια αυτά το Μαυροβούνιο συνεχίζει τι μεταρρυθμίσει του με σταθερό αριθμό. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσει να γίνει υποψήφια χώρα και θα συμφωνήσουμε τον Ιούνιο να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο. Από την πλευρά της Δανικής Προεδρίας εμείς θα συνεργαστούμε στενά με την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βάλαμη. Ακολουθεί ο κύριος Φίλε για την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Με μεγάλη χαρά και τιμή μιλώ σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συζήτηση ε, περί του ψηφίσματος για την ε, διαδικασία ένταξη του Μαυροβουνίου. Ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και τα συγχαρητήριά μου στον εισηγητή για την εξαιρετική του έκθεση. Η απόφαση του Συμβουλίου το Δεκέμβριο αναγνωρίζει την πρόοδο της χώρας τα, τελευταία, τα πέντε χρόνια μετά από την ανεξαρτησία της και ειδικότερα από το Δεκέμβριο του 2010 όπου της χορηγήθηκε το καθεστώς υποψηφίου χώρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι σε ο δρόμος για τι ενταξιακέ διαπραγματεύσεις. Κλειδί για αυτή την επιτυχία ήταν η αποφασιστικότητα των αρχών του Μαυροβουνίου να προχωρήσουν σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις με την εμπλοκή του Κοινοβουλίου, της αντιπολίτευσης, της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή η ευρεία εθνική συνένεση για την ένταξη τη χώρας στην Ευρώπη αποτελεί τεράστιο πλανέκτημα για το Μαυροβούνιο. Θα διευκολύνει τη συνεχή ομαλή της πρόοδο σταθερά προς ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνάντησα τον Πρωθυπουργό την περασμένη εβδομάδα η αποφασιστικότητά του να προχωρήσει με τις μεταρρυθμίσεις και η δέσμευσή του για διατήρηση της προόδου στο πλαίσιο της ατζέντα ε, της χώρας για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αξίζει συγχαρητήρια. Η έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης δεν θα σημάνει το τέλος της διαδικασίας, αλλά την έναρξη ενός μεγάλου και απαιτητικού ταξιδιού. Αξιότιμα μέλη, όπως αναγνωρίζετε στην εκτίση του κυρίου Τάνεκ, το Μαυροφούνιο έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο μέχρι σήμερα, αλλά θα χρειαστεί να αφιερώσει ακόμη περισσότερες προσπάθειες ε, για το κράτος δικαίου, ειδικότερα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος η έκθεση ήταν και που αφορά ε, ειδικότερα τη ε, διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να ε, εξεταστούν και να διερευνηθούν όλες οι σχετικές υποθέσεις. Σε συμφωνία με την συνένεση του 2006 για τη διεύρυνση γνωρίζουμε ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε πρώιμο στάδιο της ενταξιακής διαδικασίας. Η νέα προσέγγιση για τα κεφάλαια 23 και 24 για τη δικαιοσύνη ε, και την ασφάλεια θα τους επιτρέψει θα επιτρέψει να δοθεί επαρκής χρόνο στο Μαυροφούνιο ώστε να αποκτήσει ένα σημαντικό ιστορικό στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος καθώς εγώ σας μελώ, η πρώτη διερευνητική φάση του ελέγχου του ε, άρθρου 23 ε, λαμβάνει χώρα του 24 λαμβάνει χώρα, ενώ η διερεύνηση του άρθρου 23 έλαβε χώρα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ένα άλλο σημαντικό σημείο για το Μαυροβούνιο θα είναι η οριστικοποίηση της ε, τρέχουσας συνταγματικής μεταρρύθμισης σε συμφωνία με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας ε, σε ένα πνεύμα συνένεσης και επικοδομητικού διαλόγου με τα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Αυτό θα αποτελέσει στη βαρύ εγγύηση για την ανεξαρτησία και τη λογοδοσία του δικαστικού σώματος η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων αποτελούν επίσης πρωτοβουλίες, ειδικότερα η ελευθερία έκφρασης και η μη διακριτική μεταχείριση. Η πρόσφατη επίθεση κατά ενό δημοσιογράφου που διεξήγαγε έρευνε είναι απαράδεκτη και θα πρέπει να διερευνηθεί ενδελεχώς μαζί με παρελθούσε περιπτώσεις βίας και βανδαλισμών κατά των μεσομαζικής ενημέρωση. Περαιτέρω επίσης προσπάθειες απαιτούνται για την ενίσχυση της πολιτικής μη διακριτικής μεταχείρισης ειδικότερα σε θέματα ισότητας των φύλων και αποτελεσματικής ε, προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Γίνονται όλο και περισσότερες ε, προσπάθειες. Επίσης πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των εκτοπισμένων πληθυσμών η αντιμετώπιση αυτών των εκκρεμουσών προκλήσεων βασίζεται στο, Μοντενε, Μαυροβούνιο και στην ικανότητά του να διατηρήσει το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων και να διασφαλίσει την αποτελεσματική του υλοποίηση. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες του Μαυροβουνίου σε αυτό το δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παρέχοντας οικονομική ε, και επιβοήθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, κύριο Στάνεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Μαυροβούνιο ως υποψήφια χώρα παραμένει μία σχετικά απλή υπόθεση όσον αφορά την παρακολούθηση της πρόοδου. Και εδώ πέρα το μικρό είναι και όμορφο. Το Μαυροβούνιο έχει εργαστεί σκληρά για να εκπληρώσει τα κριτήρια και τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 7 τομείς. Δηλαδή να βελτιώσει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, ο επαγγελματισμός της διοίκησης, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ελευθερία των ΜΜΕ και συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Προσφάτως ε, εντάχθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου πέρυσι το Δεκέμβριο και οπωσδήποτε η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει το Μαυροβούνιο να οικοδομήσει μια σύγχρονη ανταγωνιστική οικονομία. Πρόκειται για ένταξή του στην παγκόσμια οικονομία. Τα βασικά κριτήρια της Κοπενχάγης που συμπεριλαμβάνουν ε, σχέσεις ε, μεταξύ των ε, διαφόρων εθνοτήτων, δικαιώματα ομοφιλοφίλων, ελευθερία και ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και των ΜΜΕ. Όλα αυτά καλύπτονται στην έκθεσή μου. Χάρη στην εξαιρετική φυσική του μορφιά παίζει σημαντικός ρόλος και ο τουρισμός και άρα προστατεύεται το περιβάλλον και είναι αυτό υψηλή προτεραιότητα όσον αφορά και την ε, κατασκευή διαφόρων φραγμάτων. Θα πρέπει επίσης η χώρα να απελευθερωθεί από την γραφειοκρατία για να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις και να προχωρήσει η ανάπτυξη και οι ξένες επενδύσεις. Το Μαυροβούνιο επίσης είναι γνωστό ως μια χώρα που προωθεί την ε, περιφερειακή συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, ε, την επίλυση των διαφορών με την Κροατία των συνοριακών διαφορών και ε, είναι πρωτοπόρο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο σε μια περιοχή που δυστυχώ έχει πολύ οργανωμένο έγκλημα. Επίση, υπέγραψε με Σερβία, Πούγδημο και Κροατία συμφωνίε έκδοση. Εν ολίγη, είναι μια θετική περίπτωση το Μαυροβούνιο και ελπίζουμε οι διαπραγματεύσει να ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2012. Ο κύριος Μίτσελ τώρα. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο και αυτή την έκθεση. Μερικέ φορέ όταν ξανακοιτάμε αυτό το κομμάτι τη ιστορία δεν θα κοιτάμε μόνο για τι οικονομικέ αταραχέ αλλά και ε, θα θυμόμαστε και το γεγονό ότι έπεσε το τείχο του Βερολίνου θαυματουργά το 1989 και εδώ είμαστε ξαφνικά με κάποια κράτη-μέλη να μιλάμε για την ένταξη του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα θαύμα. Αυτό χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή, αυτό ήταν η φιλοδοξία. Αυτό ήταν το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγχαίρω λοιπόν το Μαυροβούνιο για την πρόοδο, για τον τρόπο με τον οποίο ε, αντιμετώπισε τα ζητήματα μέχρι σήμερα. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτή προς οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα που είναι δημοκρατία και μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες της ιδιότητας μέλους. Αναφέρω αυτό το ζήτημα διότι πρόκειται για ένα δύσκολο ζήτημα για τα μικρότερα κράτη-μέλη σε κάποια βάση πάλι θα πρέπει να εξετάσουμε τα θεσμικά ζητήματα. Μπορούμε να συνεχίσουμε να διευρυνόμαστε με τον τρόπο που το πράττουμε και να έχουμε μία κομισιόν με όλο και περισσότερους επιτρόπους. Η απάντησή μου είναι ναι, διότι οι μικρές χώρες ε, βοηθούν με την υποψία τους, αλλά εάν αυτό το ζήτημα πρόκειται να αντιμετωπιστεί, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τρόπο που να μην που τα κράτη-μέλη ανεξαρτήτως μεγέθους να έχουν ισότητα. Χαιρετίζω λοιπόν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και χαίρομαι που βλέπω ότι το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζει να υπάρχει και εμβαθύνουμε και κάνουμε αυτή την Ήπειρο ένα σταθερό τόπο για το μέλλον, ένα τόπο όπου μπορούμε να διεξάγουμε τις υποθέσεις μας ε, με δικαιοσύνη σε διεθνές επίπεδο. Το ρολόι μας έχει χαλάσει. Ο κύριος Φέρμε, έχει το λόγο για δύο λεπτά. Θα χρησιμοποιήσω το δικό μου ρολόι για να σας χρονομετρήσω κύριε Φέρμε. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι μπορώ να μιλήσω στο δινεκέ, αλλά ίσως όχι. Θα ήθελα αγαπητοί συνάδελφοι να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνοκ ο οποίος ξέρει ότι έχει μια μεγάλη συνένεση που τον υποστηρίζει σε σχέση με την έκθεση αυτή. Είναι πολύ θετικό να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει ένταξης με το Μαυροβούνιο. Είναι ένα θετικό μήνυμα το οποίο μπορεί να διστείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Και σίγουρα έχουμε εξετάσει τα επιτέγματα του Μαυροβουνίου και υπάρχει μια σημαντική πρόοδος. Πρέπει να επενέσουμε το Μαυροβούνιο για την ε, δέσμευσή του στην περιφερειακή σταθερότητα και στις καλές διμερείς σχέσεις με τους ε, γείτονές του. Έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο. Έχει καταφέρει να καλύψει τις κυρίες προτεραιότητες. Βέβαια παραμένουν πολλά που πρέπει να γίνουν και οι μελλοντικέ ε, ενέργειες θα πρέπει να επιτευχθούν χάρη σε πολιτική θέληση και από την πλευρά του Μαυροβουνίου για ένα κράτος δικαίου, για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της διαφθοράς του οργανωμένου εγκλήματος, του λαθρεμπορίου. Πρέπει λοιπόν το Μαυροβούνιο να εξασφαλίσει όλα αυτά για να προχωρήσει η διαδικασία της ένταξης. Επομένως, θα πρέπει να εξασφαλίσει το Μαυροβούνιο ότι θα υπάρχει και καλύτερη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών να εξασφαλίσει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, των συλλογικών ε, διαπραγματεύσεων στον εργασιακό χώρο, να σταματήσει η βία κατά δημοσιογράφων. Και είναι ανησυχητικά τα στοιχεία που έχουμε από το Μαυροβούνιο μερικές φορές σε σχέση με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τη βία κατά των δημοσιογράφων. Και επίσης είναι πολύ ε, ανισχυτικό το ότι είναι πολύ μικρή εκπροσώπηση των γυναικών στα ανώτατα αξιώματα του Μαυροβουνίου. Θα χαιρετήσουμε ιδιαίτερα το να επιτευχθεί η εκπλήρωση των κριτηρίων από το Μαυροβούνιο και επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το πρωτεξιακό πρόγραμμα είπα, να είναι με τέτοια μορφή ώστε να μπορέσει να δώσει δυνατότητα στο Μαυροβούνιο να προσαρμοστεί το ταχύτερο δυνατό. Ο κ. Βάγκλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νόμιζα πως ε, εσείς κύριε Πρόεδρε ως φιλελεύθερος ε, θα το πως το σταματήσατε επίτηδες το ρολόι για να μιλήσουμε περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνοκ ε, για την εξαιρετική συνεργασία και όλους τους άλλους τους σκιώδεις εισηγητές. Είναι καλά αυτά τα νέα για το Μαυροβούνιο και για εμάς οι διαπραγματεύσεις ξεκινάνε τέλος Ιουνίου ή Ιούλιο. Θεωρούμε πως το Μαυροβούνιο είναι προετοιμασμένο και η συνοχή στην κοινωνία επίσης υπάρχει. Θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο θετικό είναι πως το Μαυροβούνιο ξεκινάει με ένα από τα δυσκολότερα κεφάλαια, το υπαριθμόν 23, το Μαυροβούνιο έχει περάσει πολλές δύσκολες μεταρρυθμίσεις, μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, θεσμικά όργανα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και αυτό είναι κάτι το οποίο ανέφεραν πολλοί ευρωβουλευτές. Επίσης θέλουμε να αναφέρουμε το σημαντικό ρόλο που παίζει στην περιφερειακή συνεργασία. Όπως και ο συγητής έτσι και εγώ θεωρώ πως η απόφαση να παραπευθεί το ζήτημα των συνόρων χωρικών υδάτων στην Χάγη είναι κάτι το θετικό. Καλωσορίζουμε τα βήματα που έλαβε η κυβέρνηση του Μαυρομουνίου για την ε, ελευθερία έκφρασης ε, και για την ανοχή όλων των μειονοτήτων στην ε, κοινωνία. Κάποια από αυτά τα ζητήματα είναι καινούργια για την κοινωνία του Μαυρογονίου, αλλά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχει φτάσει λοιπόν η στιγμή αυτή η μικρή αλλά πολύ όμορφη χώρα να ακολουθήσει μια ευρωπαϊκή πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ξαναλειτουργεί το χρονόμετρο. Η κυρία Λούνα Τσεκ για μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Υπουργέ Βάμεν, συνάδελφοι, ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Τένοκ για την εξαιρετική έκθεσή του και την επικοδομητική συνεργασία που μας βοήθησε να επιτύχουμε συμβιβασμούς εκ μέρους των Πρασίνων. Ήθελα επίσης να χαιρετήσω τη σαφή υποστήριξη που θα δώσει αύριο αυτό το Κοινοβούλιο για την άνοιξη των διαπραγματεύσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση με το Μαυροβούνιο. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προ τα εμπρό και έτσι θα διατηρήσουμε αυτή την ορμή διεύρυνση με την Κροατία, με την η υποψηφιότητα της Σερβίας, ε, ναι, το Μαυροβούνιο είναι έτοιμο και πάει πάλι πολύ καλά. Πολλές τροπολογίες που υποβάλαμε έγιναν δέκτες ε, ψηφίστηκαν ε, στη Σχετική Επιτροπή. Ήταν πολύ θετικό όλο αυτό, αλλά παραμένει ένα πρόβλημα στο Μαυροβούνιο η διαφθορά έχει συζητηθεί και έχει αναφερθεί από πολλούς συναδέλφους ειδικότερα όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων αλουμινίου, τηλεπικοινωνίες. Έγιναν διαδηλώσεις ε, πρόσφατα και πραγματικά η κυβέρνηση πρέπει να το φροντίσει να το αντιμετωπίσει. Επίσης, ε, οι απειλές που δεν είναι μεμονωμένες υποθέσεις ε, και η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωσης. Επίσης, ο νόμος για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, η υλοποίηση αυτού του νόμου, εκχωρείται ουσιαστικά στην εκλογική επιτροπή του κράτους και ξέρετε από ποιον αποτελείται, από εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων. Δεν είναι αυτό τρόπο για να ελέγχουμε τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Ας τελειώσω με μια θετική απόψη όσον αφορά τα ζητήματα LGBT για τους ομοφιλοφίλους. Θα ήθελα να προσθέσω μια πτυχή περιφερειακής πρωτοβουλίας στο Μαυροβούνιο και η κυβέρνηση διεξήγαγε πρόσφατα μια περιφερειακή συνεδρίαση για τους ομοφιλόφιλους με την Κροατία και αυτό είναι καλό. Κύριε Χουντή, ένα λεπτό. Τις συνάδελφοι είναι υπέρ της ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και άλλωστε όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων εφόσον ο λαός το επιθυμεί, εφόσον οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνούν. Όμως πιστεύουμε πως αυτή η διαδικασία, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να αποτελέσουν την αφορμή να λυθούν προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά, δημοκρατικά, προβλήματα δικαιωμάτων σε όφελος του λαού. Με αυτή την έννοια η έκθεση έχει τέτοιες θετικές προτροπές ιδιαίτερα στην καθιέρωση ενός σύγχρονου δημοκρατικού κράτους, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Έχει όμως δύο σημεία που με την ευκαιρία που η περίπτωση του Μαυροβουνίου είναι από τις πιο εύκολες που έχουμε στα Βαλκάνια, θα ήθελα να τα τονίσω λέγοντας ότι δεν συμφωνούμε να τίθενται, να τίθενται τέτοια ζητήματα ή με αυτόν τον τρόπο. Το πρώτο θέμα είναι ότι συμψηφίζει την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ το νατο όπω ξέρετε είναι ένα προβληματικό οργανισμό και ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή δεν έχει την καλύτερη φήμη μιλάω στην περίπτωση της γενικότερης ε, Βαλκανική και το δεύτερο σημείο έχει να κάνει ότι ουσιαστικά προτρέπουμε σε οικονομικέ λύσει, όπω α πούμε ξένε επενδύσει, ελαστικοποίηση τη εργασία, που είναι σίγουρο υπάρχει ψηλή ανεργία στο μαυροβούνιο ότι θα επιδεινώσει την κατάσταση των εργαζομένων και επομένω θα μπει αν θα μπει με τέτοια κριτήρια το μαυροβούνιο κατεβάζοντα το γενικό επίπεδο οικονομική και κοινωνική στάθμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να μην ήταν αυτά τα σημεία στην έκθεση του συναδέλφου. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Και ε, Μακοβέη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Κατά το τελευταίο έτος το Μαυροβούνιο έχει σημειώσει ε, πρόοδο όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος. Έχουν ληφθεί μέτρα ενίσχυσης της λογοδοσίας, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσμάτων των δικαστών και των εισαγγελέων. Αυτά όμως βρίσκονται μόνο σε χαρτί και σε νομοθεσία. Η υλοποίηση είναι το σημαντικότερο, είναι το ζήτημα κλειδί και είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί. Εάν κοιτάξουμε τα τελευταία 20 χρόνια σε, αυτές, σε αυτή τη χώρα, σε αυτές τις χώρες τις ε, πρώην κομμουνιστικές, οι πιο δύσκολες μεταρρυθμίσεις ήταν οι μεταρρυθμίσεις του δικαστικού σώματος και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Για την καταπολέμηση της διαφθοράς είχε ενισχυθεί η νομοθεσία με την υιοθέτηση μιας νέας νομοθεσίας για την εισαγγελία, για την ίδρυση πολιτικών κομμάτων και για τη σύγκρουση συμφερόντων. Αλλά και πάλι η εφαρμογή είναι το ζήτημα κλειδί και ε, το κλειδί για την εφαρμογή όλων αυτών θα πρέπει να διασφαλιστεί ένα προβλέψιμο δικαστικό σύστημα και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού. Η νομολογία πρέπει να ενοποιηθεί, δεν πρέπει να είναι τυχαία και όλες οι αποφάσεις πρέπει να δημοσιοποιούνται. Για την καταπολέμηση της διαφθορός, διαφθοράς οι αρχές του Μαυροβουνίου πρέπει να εστιαστούν στις περιπτώσεις υψηλή διαφθοράς. Αυτό θα αποτελέσει δοκιμή απόδειξης της αξιοπιστίας της πολιτικής τάξης και του δικαστικού σώματος. Χρειάζονται ε, οι πολίτες του Μαυροβουνίου ένα πλέον ε, διαπιστευμένο ιστορικό αντιμετώπιση των σοβαρών υποθέσεων. Κύριε Μπασέσκου, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Μαυροβούνιο έχει επιτύχει μεγάλη πρόοδο στο τελευταίο καιρό που έχουν τονιστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλω να χαιρετήσω και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε σχέση με την έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξη με τη χώρα αυτή μέσα στο 2012, τον Ιούνιο του 2012. Μπορούμε με τον τρόπο αυτό να ενθαρρύνουμε μεταρρυθμίσει σε όλε τι χώρε τη περιοχή, καταδεικνύοντα ότι οι εσωτερικέ αυτέ μεταρρυθμίσει είναι απαράγραπτο στοιχείο για να μπορέσουμε να, προωθήσουμε τη διαδικα... να προωθηθεί η διαδικασία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τι αρχέ του Μαυροβουνίου να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις του, ιδίως στον τομέα τη δικαιοσύνη του αγώνα κατά της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος. Και στο πλαίσιο αυτό Πιστεύω ότι η νέα στρατηγική της Κομισιόν για το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24 είναι ιδιαίτερα εύστοχη. Στην αρχή των διαπραγματεύσεων μάλιστα υπογραμμίζω ότι θα πρέπει όμως να υπάρξουν μέτρα τα οποία θα ληφθούν για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση των Ρωμά με μια εθνική στρατηγική για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κ. Κούκαν έχει το λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια στον κύριο Τάνοκ για τη σύνταξη της έκθεσης αλλά και για την στήριξη στην διαδικασία ένταξης του Μαυροβουνίου. Επίσης να ευχαριστήσω και τους σκιώδες εισηγητές. Το Μαυροβούνιο έχει επιτύχει αυτή η πρόοδο στα θέματα της ένταξης. Πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στο μετασχηματισμό της κοινωνίας αφορά τις πολύ γνωστές 7 προτεραιότητες ε, που έχει η Κομισιόν διαδικασίες που πρέπει να ενισχυθούν Βεβαίως ε, υπάρχουν ακόμα πολλά εκκρεμή ζητήματα όσον αφορά το κράτος δικαίου, κατά πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς, ε, συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, αλλά και σε αυτούς τους ε, τομείς υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Όλα αυτά είναι διαδικασίες οι οποίες έχει κάποια μέσα στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Μαυροβούνιο. Τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να το στηρίξουμε στις ε, προσπάθειες του. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πόσελτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Μαυροβούνιο είναι μια μια χώρα ξεκάθαρη ευρωπαϊκή, το αρχαιότερο από τα νέα κράτη στα Βαλκάνια με σλαβική και αλβανική κουλτούρα, χώρος συνάντησης μουσουλμάνων και χριστιανών. Η προστασία των μειονοτήτων είναι πάρα πολύ καλή, οπότε παρά τα προβλήματα που υπάρχουν θεωρώ πως το Μαυροβούνι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο που πρέπει να στηρίξουμε έντονα. Γι' αυτό χαιρετίζω την εξαιρετική έκθεση Τάνοκ και θεωρώ πράγματι πως ε, μαυροβούν οι βουλευτές και ε, ένας επίτροπος θα εμπλωτίσουν ε, νομίζω το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση από το Λουξεμβούργο αυτό των Βαλκανίων. Ωραία. Λέω πρώτος. Κύριε Φίλε, έχετε λόγο. κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Θέλω να ολοκληρώσω τι παρατηρήσει μου επαναλαμβάνοντα τα συγχαρητήριά μου προ τον Τσαρτσδανόκ, τον εισηγητή για την ενημερωμένη του συμβολή στη σημερινή συζήτηση. Είμαι πεπισμένο ότι αυτό το ψήφισμα στέλνει το σωστό μήνυμα στο Μαυροβούνιο. Τόσο την αναγνώριση τη σκληρή δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά και ισχυρή ενθάρρυνση για τη συνέχιση ε, της ε, διαδικασίας με αποφασιστικότητα. Βρίσκεται το Μαυροβουνίο πολύ κοντά στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και είμαι βέβαιο ότι με τη συμμετοχή του λαού του και την κοινή υποστήριξη θα αποτελέσει παράδειγμα για την περιοχή προχωρώντας στις προσπάθειες ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα τελευταία, ε, πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου, αυτή την άνοιξη η Κομισιόν θα συντάξει μια ενδιάμεση έκθεση για τα προγράμματα ε, υλοποίησης του Μαυροβουνίου και τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα, ειδικότερα για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα εξετάσει την πρόοδο όσον αφορά τις 7 προτεραιότητες ε, κλειδιά μετά από την έκθεση πρόοδου του 2011. Εφόσον ε, αποδειχθεί ότι υπήρξε πρόοδος τον Ιούνιο, θα ε, διαπιστωθεί η εξοπιστία της διαδικασίας διεύρυνσης. Για το Συμβούλιο, κύριε Υπουργό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί βουλευτές, οι πολίτες του Μαυροβουνίου έχουν μια ελπίδα. Η ελπίδα τους αυτή είναι το μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μια απτή και εφικτή ελπίδα. Το Μαυροβούνιο έχει μια εθνική ενότητα σε σχέση με το θέμα της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε λοιπόν πόσο γρήγορα έχουν αρχίσει να πραγματοποιούνται αυτές οι ελπίδες. 21 Φεβρουαρίου εφέτος πήγα στο Μαυροβούνιο και είδα μια θέληση για μεταρρύθμιση και μια στεναρή δέσμευση από τις πολιτικές ελίτ. Μέσα σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έγιναν σημαντικές μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση ενός κράτους δικαίου το οποίο θα μπορεί να εγγυάται για τα βασικά δικαιώματα των πολιτών. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, παραμένει ακόμα να επιτευχθούν πρόοδοι σε πολλούς τομείς, κυρίως σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Στα πλαίσια αυτά, εγώ περιμένω την επόμενη έκθεση προόδου της Κομισιόν για την αξιολόγηση των ενεξελίξη ενεργειών μεταρρύθμισης. Έχουμε αναφέρει σήμερα πολύ σημαντικές ανάγκες για μεταρρυθμίσεις και υπάρχει συνένεση μεταξύ Μαυροβουνίου και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τους τομείς όπου πρέπει να επέλθει πρόοδος. Πάνω απ' όλα το Μαυροβούνιο θα πρέπει να εστιάσει στην συνταγματική μεταρρύθμιση και μέσω αυτής την αντιμετώπιση της διαφθοράς του οργανωμένου εγκλήματος και την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας. Επίσης το θέμα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και η νομοθεσία κατά των διακρίσεων πρέπει να βελτιωθούν. Εμείς θα παρακολουθήσουμε λοιπόν και τις ενέργειες σε σχέση με την σύνταξη του νέου συντάγματος γιατί πρέπει να εξασφαλίσουν και την ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου. Υπάρχουν λοιπόν μία σειρά από αιτήσει, όπως παραγωγή χάρη ένα του Μαυροβουνίου, ενίσχυση της ε, ε, αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και όλα αυτά έχουν αποφέρει και καρπούς Φυσικά το Μαυροβούνιο έχει αντιμετωπίσει και την οικονομική κρίση και η οικονομία του Μαυροβουνίου θα πρέπει να μπορέσει να αναπτυχθεί περισσότερο και αυτό σημαίνει ένα, έφορο, ένα πιο έφορο κλίμα για τη λειτουργία των επιχειρήσεων είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί μια λειτουργούσα οικονομία της αγοράς, κάτι το οποίο υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι σίγουρο όμως ότι τα πράξει αυτά το Μαυροβούνιο, θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας ε, Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Νομίζω ότι η διαδικασία ένταξης του Μαυροβουνίου αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από τα επιτεύγματα του Μαυροβουνίου. Αυτό είναι θετικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί και η διαδικασία του Μαυροβουνίου ε, θα εμπνεύσει και άλλες χώρες της περιοχής να ακολουθήσουν την ίδια κατεύθυνση. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε βάσει της έκθεσης προόδου της Κομισιόν να συνιστήσουμε την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο τον Ιούνιο του 2012. Όλα αυτά είναι προφανώς προς το συμφέρον του Μαυροβουνίου, αλλά θα προτρέψουν και άλλα κράτη των Δυτικών Βαλκανιών να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τους δώσει μια περαιτέρω όθηση. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό και για το Μαυροβούνιο και για τα, και για τα Βαλκάνια, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει περαιτέρω πρόεδρος και η Κομισιόν μαζί με το Κοινοβούλιο θα και η Προεδρία τη Δανική θα εργαστούν για να υπάρξει περαιτέρω πρόοδο και θετική απόλυξη της διαδικασίας για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 11.30. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Περνάμε τώρα